Bien, mesdames, messieurs, gagnez vos places, s'il vous plaît. Κυρίες και κύριοι, Γαλιλαίος Ψιν, ο κύριος Κέλμελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε λίγο αργήσει και για να μην καθυστερήσουμε άλλο, να προτείνω να δούμε αν μπορούμε κάποιες ε, ψηφοφορίες να τις δούμε από κοινού, κάποιες τροπολογίες να, βάλουμε συν σε κάποιες από κοινού για να μην χάνουμε χρόνο και τις ψηφίζουμε όλες μία-μία. Σας ευχαριστώ για αυτή τη διευκρίνηση κύριε Κιόλμερ. Καταρχάς, να βεβαιωθώ ότι έχετε μαζί σας τις κάρτες ψηφοφορίας. Τις έχετε βάλει στα ηλεκτρονικά μηχανήματα. Άρχεται η ψηφοφορία. Δοκιμή κάνουμε. Δοκιμή είναι όχι ψηφοφορία. Λείπουν δύο. Συνάδελφοι που έβαλαν τις κάρτες τους στο μηχάνημα αλλά δεν ψηφίσαν Τρεις τώρα. Δύο, βάλατε την κάρτα σας στο μηχάνημα αλλά δεν ψηφίσατε. Εγώ αυτή τη φορά ψήφισα. ένα τώρα. Μία τέλος πάντων. Πέρας. Πρέπει καταρχάς να ακούσουμε τον κύριο Γκέγερ. Για τρεις μεταφορές που αφορούν τον προυφολογισμο 2017 τμήμα 3. Κύριε Γενική Συγητά, ανακεφαλαίωση μπορούμε να τα ψηφίσουμε και τα τρία μαζί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, έχουμε τρεις διαφορετικές μεταφορές κονδυλίων και διαφορετικές και σε όγκο. 12. Η 12 έχει να κάνει με το διοικητικό προπολογισμό. Η Κομισιόν ζητά τα μέσα γιατί ο Ευρωπαϊκό Σχολείο στη Φραγκφούρτη για με 4,6 εκατομμύρια να τα πάρουμε από το διοικητικό απόθεμα. Ο λόγο είναι ότι η διαπραγματεύσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Κομισιόν για το κόστο και τη συμμετοχή στο κόστο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί επιτυχώ, οπότε μπορούμε να δούμε γιατί και πότε θα γίνει η ολοκλήρωση. Οι άλλες δύο κατηγορίες έχουν να κάνουν με την κατηγορία 4, εξωτερική πολιτική. Από τη μία έχουμε μεταφορά 13 εκατομμυρίων ευρώ από το μέσο για τη σταθερότητα και την ειρήνη που πάνε στο, Ευρωπαϊκό, στο μέσο Ευρωπαϊκής Γειτονίας για να πρικοδοτηθεί το Ταμείο για την Αφρική και η άλλη μεταφορά είναι στην κατηγορία πάλι 4. Η 3, μιλάμε για ένα μεγάλο ποζό, 184 εκατομμύρια υποχρεώσεις και 130 πληρωμές ζητούνται για την ενίσχυση ανθρωπιστικής βοήθειας από, την, ε, από το απόθεμα επίγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση ε, ε, καταστροφών στο κέρας της Αφρικής. Όχι για να τις αποφύγουμε, αλλά τέλο πάντων για να μειώσουμε τον αντίκτυπό τους. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και για τα τρία. Έχω ένα ερώτημα για την Κομισιόν, ωστόσο. Η μεταφορά 15, 16, 17 από δύο διαφορετικές πηγές έχουν πάρθει τα ποσά αυτά. Για το 16 και το 17 όμως είναι τα ίδια. Καλή, είναι, έρχονται από το 14.02.42 για το απόθεμα δηλαδή το, α, για τις επίγουσες ανάγκες και πάνε πάλι στο απόθεμα για τις επίγουσες ανάγκες. Πώς δεν, δεν θα ήταν καλύτερο ή πιο εύκολο να τα κάνουμε αυτά τα δύο ένα αφού είναι τα ίδια. Μάλιστα, για αυτές τις μεταφορές να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, κύριε Γκάγερ. Ναι, να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Συμφωνεί και η Επιτροπή. Όχι, δεν συμφωνείτε. Για την πρώτη μεταφορά. Έχετε κάτι να απαντήσετε κύριε από την Επιτροπή στην ερώτηση του κυρίου Γκάγερ. Ναι, πολύ γρήγορα για να απαντήσω στον κύριο Γκάγερ. Η ερώτηση είναι γιατί έχουμε διαφορετικές προτάσεις μεταφορών για αυτές τις τρεις κρίσεις. Είναι απέτηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Για κάθε κρίση να υπάρχει ξεχωριστή πρόταση για μεταφορά από τη Δημοσιονομική Αρχή. Λέω θα πηγαίνανε σε μία. Το ερώτημα είναι 15, 16, 17. Σχετίζονται με την ίδια κρίση, ανθρωπιστική κρίση στο κέρας της Αφρικής. Παίρνετε τα λεφτά από δύο διαφορετικές πηγές. Μία από το, ε, τις επίγουσες ανάγκες, το αποθεματικό για τις επίγουσες ανάγκες και μία από το είναι προταξιακή βοήθεια. Αυτή από τις επίγουσες ανάγκες έχει, έχει χωριστεί σε δύο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν θέλω να καθυστερήσουμε τη διαδικασία. Απλώς για να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται ρωτώ. Um, Υπάρχουν τρεις μεταφορές γιατί είναι τρεις διαφορετικές κρίσεις. Η μία είναι το κέρα της Αφρικής, η δεύτερη είναι το Ιράκ, η δεύτερη μεταφορά και η τρίτη η Συρία. Ίσως η σύγχυση προκύπτει διότι υπάρχει ένα μικρό ποσό επαναχρησιμοποίησης που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την προενταξιακή βοήθεια για μια από τις μεταφορές. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε λοιπόν μεταφορά 12. Ελεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. «26 υπέρ 3 κατά εγκρίνεται η μεταφορά». Τώρα, μεταφορά 14-2017. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 22 προς 4, δύο εποχές. Μεταφορά 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 26 προς 1 και μια εποχή. 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. 27 υπέρ, ε, μία εποχή. Και τέλος 17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, μία εποχή. Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Τάραντ για τα υπόλοιπα τμήματα και για επτά μεταφορές που δεν χρειάζεται όμως να ψηφίσουμε απαραίτητος λόγω του ποσού. Κύριε Τάραντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχει πολλές μεταφορές ακόμα, αλλά να τονίσω την πρόσφατη εμπειρία μας από τις μεταφορές. Ο προπολογισμό είναι κάτι παραπάνω από μια εκτίμηση. Είναι μια πρόβλεψη για το τι μπορεί να γίνει και πολλές φορές περιλαμβάνει προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα. Ο προπολογισμό όμως ε, καταγράφει και μια δέσμευση ε, σε σχέση με τις προβλέψεις για μια συμφωνία σε σχέση με το προβλεπόμενο αποτέλεσμα. Είναι ένα φιλοσοφικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει η Επιτροπή μας. Και για να σας δώσω και μια ιδέα για τις σημαντικές αλλαγές που επιφέρονται από τη δράση του ηλεκτρικού συνεδρίου και τις δαπάνες του. Το σύνολο των μεταφορών αυτών είναι 476 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 45 πηγαίνουν στην ψυχαγωγία και τις δαπάνες εκπροσώπησης για τα μέλη των θεσμικών οργάνων Δύο είναι για τους εορτασμούς του, ε, της επαιτίου του δικαστηρίου. Της 40ης επαιτίου η οποία το, ε, όταν συμφωνήθηκε δεν ε, είχε προβλεφθεί στον προπολογισμό. Όμως η εκλογή του Εστονού ε, ελεγκτή οδήγησε στον αποφασιστή να ε, εορταστεί αυτή η επέτειος. Οι Εστονοί αρέσκονται στα πάρτι. 60.000 ε, επίσης για την ε, κάλυψη των παιδικών σταθμών του ελεγκτικού συνεδρίου, 25.000 για τις αλλαγές στο, στην εστίαση. τα οποία τα υπόλοιπα θα μπορούσα να τα δω και θετικά και να ζητήσω από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν αυτές τις μεταφορές. Ευχαριστώ. Το μικρόφωνο σας, Πρόεδρε. Ναι, άρα επτά μεταφορές προτείνεται να εγκρίνουμε. Ποιε μεταφορέ δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε επισήμω λόγω του ποσού. Α τα εγκρίνουμε όλα μαζί. Να τα εγκρίνουμε ε, βάσει των όσων μα είπε ο εισηγητή. Να, θεωρώ ότι, να θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Όχι, θέλετε ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν θα ψηφίσουμε. Να τα ψηφίσουμε αν μπλοκ. Κύριε Φίντ, δέχεστε. Θα έφερνα αντίρρηση και θα προτιμούσα να τα ψηφίσουμε ξεχωριστά παρόλο που ήθεστε, ήθιστε. Εσείς αποφασίζετε, εσείς είστε ο πρόεδρος, θα ακολουθήσω την προτροπή σας. Εγώ θέλω να διευθύνω τις συζητήσεις και να επιτρέψω να εκφραστεί ποικιλομορφία. Είμαστε σε ένα θεσμικό όργανο βαθιά δημοκρατικό. Δεν θέλω να βγείτε αυτή την αίθουσα απόψε με ματαιώσεις και απογοητεύσεις. Ας τοποθετηθούμε για την πρώτη από αυτές τις μεταφορές. 0317 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται 24 προς 3. 04 Α, 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Όχι, αλλά η ψηφοφορία έληξε. 22 υπέρ 3 κατά. α 17 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 υπέρ 3 κατά. 07C17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 υπέρ 3 κατά. 08 17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 24 υπέρ 3 κατά. 08 μόλις το είδαμε. Δεν ψηφίσαμε το 05C17. Άρχεται η ψηφοφορία. 05C17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 24 προς 3. Και τέλος 09C17 άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες όχι. Πέρας. 21 υπέρ 3 κατά. Πολύ ωραία. Περνάμε στις πιστώσεις των κτηρίων. Έκθεση Χόλμαγερ. Ο κύριος Τάραντ μας είχε πει για δύο μεταφορές που έφτασαν αργά στην Επιτροπή μας, οπότε σε κάθε περίπτωση θα ψηφίσουμε στις 30 και 31 Αυγούστου. Θέλω να τις παρουσιάσετε παρόλα αυτά, ο λόγος εσάς κύριε Τάραντ. Εάν λέτε να ψηφίσουμε 31 Αυγούστου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Φτάνει με το δύσκολο σημερινό τοπίο με τις μεταφορές, διότι το ελεγκτικό συνέδριο ήταν ήδη βαρύ θέμα και ο Χέλμερ Μπρόκ ήταν εδώ από τότε που γεννήθηκε. Και θα ψηφίσουμε πράγματα ηλικίας 20 ετών. Οπότε καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που ψηφίσαμε προς στιγμή. Non, nous, nous resterons là, puisque de toute façon, le Κοιτάξτε, έτσι και αλλιώς η ψηφοφορία θα γίνει στις 30 ή στις 31 Αυγούστου. Τώρα θα αναφερθούμε στην κτηριακή πολιτική. Δύο δράσεις. Η πρώτη αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αγορά κτηρίου για την αντιπροσωπεία στην Κολομβία και θα υπάρξει συνεργασία με την Φιλανδία. Λοιπόν, η συγγήτρια είναι υπέρ, δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, τη θέτω σε ψηφοφορία την πρόταση αυτή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίζεται. πέρα της ψηφοφορίας. 21 υπέρ, 2 κατά, 2 εποχές. Η δεύτερη δράση είναι αγορά κτηρίου στην Κάνα, με, με την Γερμανία θα συνεργαστούμε για την εκμετάλλευση του κτηρίου. Ψηφίζουμε. Τέλος. 23 υπέρ, 3 κατά. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να ελέγξω το χρόνο. Χρειάστηκε ε, περισσότερος χρόνος. Ήταν ενδιαφέροντα τα θέματα. Δεν υπάρχουν στα διάφορα κάποιες παρατηρήσεις. Οι επόμενες συναντήσεις μας προβλέπονται την 30η και 31η Αυγούστου και 14η Σεπτεμβρίου. Καλές διακοπές. Υπότιτλοι AUTHORWAVE